και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με τη συζήτηση για το 2030 να επανέλθουμε και στα πιο δομικά προβλήματα που συνδέονται με το σύστημα. Ευχαριστώ κυρία Ελκάρτ. Κλείνει η συζήτηση λοιπόν. Ακολουθεί κατόπιν η συζήτηση για τους επιτρεπόμενους χειρισμούς υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα. Ο εισηγητής δεν θα μιλήσει. Ξεκινάνε οι μιλητές εξ των ομάδων. Ε, κυρία Ζόμαρη, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κανονισμός του 2006 για τους χειρισμούς υγείας είναι μια ιστορία ατελείωτη. Δεν εφαρμόζεται. Λείπουν τα διατροφικά προφίλ. Γιατί, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφαρμόσιμο επιστημονικά. Εμείς το λέμε, το έχουν πει πάρα πολύ στο Κοινοβούλιο, αλλά τελικά αποφασίστηκε να μπουν αυτά τα διατροφικά προφίλ. Γιατί δεν λειτουργούν όμως αυτά. Δεν μπορούμε να κατατάξουμε τα τρόφιμα σε καλά και κακά. Υπάρχουν μόνο καλά και λιγότερο καλά. Και βεβαίως κανείς δεν ζει ολόκληρη μέρα από ένα μόνο τρόφιμο. Οπότε δεν έχει νόημα να αξιολογήσουμε ένα τρόφιμο μεμονωμένο. Αυτά τα λέγαμε πάντα οι χριστιανοδημοκράτες του ΕΛΚ. Τώρα η Κομισιόν θέλει να εισαγάγει αυθαίρετα ένα κριτήριο για τα προφίλ αυτά για να επανέλθει δηλαδή από την πίσω πόρτα διατροφικό προφίλ για μεμονωμένα προϊόντα γιατί βεβαίω, όταν μιλάμε για την αξιολόγηση ζάχαρη, de facto έχουμε ένα διατροφικό προφίλ. Εδώ πέρα όμως παραβαίνει την νομοθεσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού. Η αντίρρησή μου απέναντι στην ε, πρόταση της ε, Κομισιόν είναι λοιπόν αντίρρηση αρχής, γιατί δεν είναι δυνατόν από την πίσω πόρτα ε, κάθε φορά να προσπαθεί να εισαχθεί ε, προφίλ διατροφικό για το κάθε ξεχωριστό προϊόν. Όχι, θα είναι ανακατηγορία προϊόντων. Να εφαρμόσει η Κομισιόν αυτά τα οποία ισχύουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχει αντίστοιχη άποψη και από το Συμβούλιο και από την ΕΦΣΑ. Και λένε, οι ίδιοι οι υπάλληλοι της Κομισιόν δεν μας ενδιαφέρει τι λένε οι επιστήμονες, εμείς το θέμε γιατί το θέμε. Δεν είναι δυνατόν. Και δεν είναι δυνατόν βεβαίω να πουλάμε διαφήμιση έτσι. Σα ευχαριστώ κυρία Σχαλτεμόζε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ομάδα του ΕΛΚ, η κυρία Σόμερ, θέλει να σταματήσουν οι διατροφικοί ισχυρισμοί διότι θεωρεί ότι δεν μας επιτρέπουν να μπορούμε να ζήσουμε μια καλή ζωή. Θέλουμε να έχουμε ισχυρισμού για τη διατροφή, αλλά αν ακούσουμε αυτά που λέει ε, το ΕΛΚ, θα φτάσουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. το διατροφικό αυτό προφίλ θα ισχύει για όλα τα τρόφιμα, για ε, πλάκες σοκολάτας, ε, για οτιδήποτε. Και τελικά στα σούπερ μάρκετ απλώς θα έχουμε δηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, η σοκολάτα κάνει καλό στο μυαλό. Ε, και αυτό τι γίνεται, ε, ευνοεί τις πολυεθνικές όπως την Εστλέ και όλες τις υπόλοιπες οι οποίες <coughs> κατακλείζουν τα σούπερ μάρκετ. Ο μόνος τρόπος λοιπόν ο οποίος έχουμε για να αποφύγουμε αυτοί οι ισχυρισμοί ε, να ξεφύγουν τελείως από τα όρια είναι να υποστηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έχει σήμερα. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να μειώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται αυτοί οι εγκεκριμένοι ισχυρισμοί και θέλει να μην μπορούν να μπουν αυτοί οι ισχυρισμοί σε κάποια προϊόντα τα οποία ε, θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα. Ζάχαρη, ε, γλυκαντικές ουσίες, ε, γλυκά και το καθεξής. Και αυτό φυσικά αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης ή η σκλήνηση κατά πλάκας ε, θα πρέπει ε, να μπορούμε να, το, να μην εφαρμόζουμε αυτούς τους ισχυρισμούς. Θα πρέπει να δίνονται στους καταναλωτές μια πραγματική εικόνα ε, για το τι συνεισφέρει στην υγεία τους και τι όχι. Είμαστε λοιπόν κατά της άποψης του ΕΛΚ να απορρίψουμε την πρόταση για τους ισχυρισμούς και είμαστε υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Σάλντε Μόσερ. Ο κύριος Σλέιτερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, η Κομισιόν έχει καταθέσει μια πρόταση η οποία δεν περιλαμβάνει αρκετούς περιορισμούς και απλώς κάνει πιο δύσκολη τη διαδικασία. Το ερώτημα μου όμως είναι το εξή. Τι θα γίνει με τα κράτη-μέλη. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα είχαν, είχαν ποτέ τη δυνατότητα να πούν όχι σε αυτή την πρόταση. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια πλειοψηφία 100 μελών που θεωρεί παράξενο όταν αγοράζει κανείς ε, μακαρόνια να υπάρχει ένα κείμενο που να λέει πώς το να τρώει κανείς δατάθρακες μπορεί να βοηθήσει το μυαλό τους. Υπάρχουν ε, τώρα άτομα τα οποία πλήττονται επειδή δεν τρώνε αρκετά μακαρονιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έχω αμφιβολίες. Εγώ νομίζω ότι η Κομισιό λοιπόν και το Συμβουλίο θα πρέπει να επομιστούν τις ευθύνες τους και να πούν κάτι το οποίο είναι αληθές, μπορεί να είναι αληθές, αλλά δεν έχει θέση στις συσκευασίες των τροφίμων. Αλλά τώρα μόνο εμείς σαν καταναλωτές μπορούμε να διαλέξουμε θα αγοράσουμε το ένα ή το β προϊόν. Αλλά για τις ταμπλέτες δεξτρόζης, για τα τρόφιμα που έχουν ζάχαρη, ε, θα πρέπει να υπάρχει παντού μία ε, ετικέτα και μία εξαίρεση. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα να λέγαμε όχι για να μην υπάρχει καμία απολύτως παροχή αυτών των πληροφοριών. Κανείς δεν ξέρει λοιπόν πού θα μπορούσε να καταλήξει μια τέτοια διαδικασία. Θα μπορεί σε όλο και πιο παράλογα προϊόντα να υπάρχουν επιγραφές και μηνύματα τα οποία λένε για τη διατροφική τους αξία. Υπάρχει λοιπόν μια πλειοψηφία πιστεύω και στους πληθυσμούς μας και στις κυβερνήσεις μας αν μας ρωτούσε κανείς που θα λέγανε ας σταματήσουμε να έχουμε αυτούς τους γελίους ισχυρισμούς και τις ταμπέλες στα τρόφιμά μας. Οι καταναλωτές μπορούν να καταλάβουν πράγματα τα οποία έχουν λογική και σχετίζονται με τα θέματα αυτά, αλλά κανείς δεν πλήττεται από την ελψίδα των θράκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Σλίτερ. Τελείωσαν οι ομιλητέ. Περνάμε εξ των ομάδων. Περνάμε στην οφθαλμοσυλληπτική διαδικασία με την κυρία Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, να πω ότι αυτή η συζήτηση πραγματικά μου κόβει την όρεξη. Αν καταφέρουμε να φάμε βέβαια και βραδινό απόψε, διότι αναφερόμαστε σε ισχυρισμού οι οποίοι προκαλούν σύγχυση στου καταναλωτέ. Και συμφωνώ με τον προναλήσαντα. Δεν θέλουμε παραπλανητικούς ισχυρισμού και γελίου ισχυρισμού στα τρόφιμα και πολλέ φορέ είναι γελοί ισχυρισμοί. Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες ε, τελούν όλο και περισσότερο υποσύγχυση. Παρά του ισχυρισμού που υποτίθεται ότι διευκρινίζουν τα πράγματα, ε, δεν ε, καταφέρνουν να κατανοήσουν ποια είναι πιο εύκολη διατροφή. Και όταν λέγεται για κάτι ότι είναι καλό τρόφιμο, φαίνεται ότι οι άνθρωποι προτιμούν αυτό και όχι κάποιο άλλο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν. Οι ισχυρισμοί θα πρέπει να είναι σαφεί και θα πρέπει να ακολουθούμε τι συμβουλέ των γιαγιάδων μα. Λίγο απ' όλα είναι καλό και ποικιλία είναι το άλλα στη ζωή. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν θα πρέπει τα πάντα να τα βασίζουμε σε αυτή τη βασική αρχή. Ευχαριστώ κύριε Μακίνες. Για να κλείσει η διαδικασία η, η κυρία... Κυρία Κάντενμπαχ, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω το γιατί εισήχθη αυτός ο κανονισμός. Δεν θέλουμε να μπερδέψουμε τους καταναλωτές, απλά να έχουν κάποια ασφάλεια. ειδικά όταν πρόκειται για κάποια προϊόντα τα οποία αποδεδειγμένα έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία. Αυτό είχα να πω. Σας ευχαριστώ κυρία Κάντμπαχ για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Η κυρία Χέντεγκάρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Εξότιμα μέλη. Εξ ονόματος του Επιτρόπου Μπόρκ θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να περιοριστεί η χρήση ε, ενό ισχυρισμού για την υγεία, για του υδατάνθρακε και για το γεγονό ότι υποτίθεται ότι μπορεί να διατηρήσει την καλή λειτουργία του εγκεφάλου, διότι πολλά τρόφιμα περιλαμβάνουν περίπλοκου υδατάνθρακε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται ο ισχυρισμό ε, παρά μόνο σε τρόφιμα τα οποία είναι πολύ χαμηλά σε σάκχαρα και προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν φυσικά σάκχαρα, όπω για παράδειγμα φρούτα, χυμή και δεν θα πρέπει να εμφανίζεται στην ετικέτα ενός πακέτου ζάχαρης ή και σε προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν πρόσθετη ζάχαρη όπως για παράδειγμα γλυκά, ε, ανθρακούχα ποτά και ούτε καθεξής. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν ισχυρισμοί για την υγεία πρέπει να σας πω ότι εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην αγορά χωρίς κανένα περιορισμό για την περιεκτικότητα σε ζάχαρα των ε, τροφίμων που φέρουν αυτή την ετικέτα. Και εάν συνεχιστεί θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν αυτόν τον ισχυρισμό εκτός αν υπάρξει τελική απόφαση από τους νομοθέτες. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ σημαντικό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιοριστεί ο ισχυρισμός αυτός θα πρέπει να υποστηριχθεί από εσά. Επίσης, ε, θεωρείται ότι ο ισχυρισμό θα πρέπει να εγκρίνεται μετά από πολύ αυστηρού ελέγχου και επί τη βάση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και αρμοδίων αρχών για διατροφικέ συνήθειε. Οι προϋποθέσεις χρήσης του συγκεκριμένου εγχειρισμού έχουν συζητηθεί εκτεταμένα με τα κράτη-μέλη και έχουν ε, εγκριθεί σχεδόν ομόφωνα. Το να υπάρχει ο ισχυρισμός αυτό σε προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν πρόσθετα σάκχαρα θα δημιουργήσει ε, ένα φαινόμενο ντόμινο για αυτά τα προϊόντα και ε, μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα στις συγκεκριμένες διατροφικές στρατηγικές που ακολουθούνται. Αυτή τη στιγμή η πρόταση που έχουμε αναχείραση είναι ασαφής ε, και επειδή δημιουργείται πόλωση θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αρκετοί ευρωβουλευτέ υποστήριξαν το ψήφισμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, αλλά κάποιοι είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβαίνει τι κατεξουσιοδότη συναρμοδιότητε που τις γίνονται και ζητούν να μην υπάρχει κανένα περιορισμό για το συγκεκριμένο ισχυρισμό και ε, έτσι θα μπορεί να χρησιμοποιείται ο ισχυρισμό αυτό για προϊόντα τα, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις μορφέ ανθράκων και ε, ε, πρόσθετα σάχαρα. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι άλλοι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτό ο ισχυρισμό είναι παραπλανητικός και αμφίσιμο για του ε, καταναλωτέ, διότι προωθεί τη χρήση ζάχαρη και επομένω θα πρέπει να απαγορευτεί ο συγκεκριμένο ισχυρισμό. Κάποιοι ζητούν απαγόρευση και για όλα τα προϊόντα. Σε περίπτωση που εγκριθεί το ψήφισμα από το Κοινοβούλιο, ο κανονισμός ο οποίος επιτρέπει τη χρήση του ισχυρισμού υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα εγκριθεί και ο ισχυρισμό θα παραμείνει στις αγορές. Χωρί να υπάρχει κανένα περιορισμό για την περιεκτικότητα σε σάκχαρα τροφίμων ε, που φέρουν το συγκεκριμένο ισχυρισμό και τη συγκεκριμένη ετικέτα. Γι' αυτό ακριβώ ο επίτροπο Μπόρκ και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να σα ζητήσουν να μην υποστηρίξετε το ψήφισμα αυτό, διότι αν το εγκρίνετε θα επιτρέπετε να χρησιμοποιείτε ακόμα αυτό ο ψευδής ισχυρισμό. Ευχαριστώ κύριε Χέντεγκαρτ. το ψήφισμα το οποίο θα κλείσει τη συζήτηση έχει κατατεθεί, που θα κλείσει τη συζήτηση έχει κατατεθεί από την ε, Επιτροπή